Prego. Please, can you sit? Se siamo pronti chiederei di accomodarvi ai collaboratori. Please, sit down, please. Se... Καθίστε παρακαλώ, αν είσαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την πρωινή ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Πριν αρχίσουμε τις ψηφορίες θα πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ ως εισηγητής που είναι επέλεξε να τον διδεχθώ εγώ εδώ στην ε, Προεδρία κατά την ψήφιση της έκθεσής του. Για να κάνουμε πρώτα πρώτα μια δοκιμή να δούμε αν ε, λειτουργεί η συσκευή για την ηλική ψηφοφορία και έτσι ταυτόχρονα θα δούμε. Εάν έχουμε πλήρη σύνθεση στις ε, αντιπροσωπείες των πολιτικών ομάδων ή αν υπάρχει ε, κάποιος παραπάνω ψηφίζουμε επομένως ποιος Λοιπόν, άπνα, η δική μου κάρτα δεν δουλεύει. Λοιπόν, ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το σύστημα λειτουργεί. Όλα καλά. Οπότε προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Jetzt ε, heben Okay. Jetzt Assicuriamo il collega che il suo voto sarà conteggiato a parte perché senza scarsa di voto tutti gli altri. Α, δεν είχε ψηφοφορία, οπότε θα μετρήσει χωριστά η ψήφο του. Οπότε έχουμε την πρώτη εκτέλεση τώρα, η οποία αφορά τι συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγματεύσει τη ονομαζόμενη TTIP. Πρώτη συμβεστική. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι σημειώστε την ε, ψήφο του συναδέλφου τώρα πάμε στη δεύτερη συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 12 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον ε, εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο για το 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπερθυμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, παραλείψαμε το 34. Το 31 ε, απορρίφθηκε, αλλά θα πρέπει να γίνει ψήφιση για το 34. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι εγκρίνεται, διορθώνει ο γραμματές. Α, συμπαθάτε με λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία υπερθυμών 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτο. 42. Υπέρ. Scusate, emendamento 42, si Το 42 ως προσθήκη. Chi a favore? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν, δεν μπορώ να δω όλα τα χέρια. Ε, 42 επομένω ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Πέρας. Ισοψηφία και Απορρίπτεται. Πενήντα τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Για το 57 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική παρθμόν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και πάμε τώρα στο 96, συμβαστική 96 ως προσθήκη. Τροπολογία, τροπολογία 96 ως προσθήκη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 110. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τοπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος 114 δηλαδή υπέρ. Ψηφίζουμε τώρα με το 114. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απολύπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. 115. Υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτονται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 6 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε την τροπολογία 119 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να κάνουμε έλεγχο και ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Κανοποιημένος. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πρώτος. Όχι. 111 διορθώνει πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική υπερθυμόν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στο 146 ως ε, προσθήκη στην συμβαστική Παρτιμόνιπτα 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 153 λέει ο πρόεδρος 153 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα πέρας εγκρίνεται εγκρίνεται έκανε λάθος συμπαράτημα 154. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 156, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 157, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Το πολύ 158, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το πολύ 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η Ηλεκτρός έλεγχος για το 159 ψηφίζουμε. Aperta. κιούζα. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική υπερθμών 8. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά αποχές Ευρωσέλγος για το 165 λέει τώρα η πρόεδρος. Ψηφίζουμε τώρα 165. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολία 167. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 176. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. 184 υπέρ κατά σε έλεγχος για το 184 ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη ψηφοφορίας πέρας ε, Συμβιβαστική υπαρθυμόν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το 188 θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία έλεγχο ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 195 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αν θέλετε όμως να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 203 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα φιούζω. Πέρας. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτονται. κοινή ψηφορία 204 για 205 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 206 υπέρ κατά άποχες Απορρίπτονται. για το 206 ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε πέρας Εγκρίνεται. 208. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 212. Υπέρ. Να έχετε το λόγο. Κύριος Φόξ. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο το 208 γιατί ε, εμείς ψηφίσαμε διαφορετικά. 208. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα το 208. Ψηφίσατε όλοι πέρας και απορρίπτεται. Συμπαθάτε με, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στα αποτέλεσμα των ψήφων, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια σύγχυση. 2-12. 212 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό να μην υπάρχει πρόβλημα για το 212. Ηλεκτρονική ψηφορία ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι. Συμπαθάτε με. Απορρίπτεται. 213. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές. το λοιπόν, έχουμε για το 215. Λειτουργική ψηφόρια, Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθυμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπάρχει μόνο 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ονομαστική ψηφοφορία. Είπατε, ε, ψηφίζουμε.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 Τρίτη ψηφοφορία. Προφέρει ερώτηση όσον αφορά την υπηρεσία Acer για τους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό είναι του Πρόεδρου Μπούζο. Και εδώ θέλουμε νομική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. La votazione è chiusa. ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Σιλικιώτη. Επένδυση για την πράσινη ανάπτυξη και την πράσινη απασχόληση. Έχετε το κείμενο. Συμβαστική παρτιμόν 1. Votazione compromesso 1, chi a favore? Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 8. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 ηλεκτρονικός έλεγχος για το 14. επαλήθηση. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και έγκρι. Τροπολογική υπερχόν 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εάν θέλετε, κάνουμε επαλήθευση για το 15. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Και εγκρίνεται. Δεκαέξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα. Επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε επαλήθευση ηλεκτρονική για το 20 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2, όπως ξέρετε, έχει μια εκδοχή η οποία Χθε το βράδυ συνετάχθη. Όμως έχετε λάβει το καινούργιο κείμενο. Αλλά πάμε στο 35. Καταβίπτουν οι άλλες. Τι είναι υπέρ. 35. Κατά. Απορρίπτεται. 3. Σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Αποχές. Θα γίνει επαλήθευση όσον αφορά το 48. Ψηφίζουμε, πέρας και απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Πέρασε ψηφορία. Εγκρίνεται. Το υπαριθμών 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτω. 53 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική παραθυμόν 4 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβαστική υπερθυμόν 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμόν 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφορία. Για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής υπερθμών 6. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Απερίφθη. Και τώρα. Πάμε στο 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Για το 86 θέλετε επαλήθευση. Ψηφίζουμε επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και είμαστε στο 87. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήψη για το 87. Ψηφίζουν. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 έχει αποσυρθεί. Το 90 δεν τελέσει. Συμπαθάτε με το 89 τώρα. Υπέρ. Κατά. απορρίπτονται. Απεσύρθη το υπαριθμόν 90. Το ψηφίσαμε την 89 και πάμε στο 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Λειτουργικό σύνολο για το 92. Ψηφίζουμε. Ένας ψήφος παραπάνω. Μια ψήφος παραπάνω για το ε, σοσιαλιστές. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε.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 Και τώρα πάμε στην έκθεση Γκίρεκ. Παρακαλώ προσέξτε όσο μπορείτε γιατί εδώ είναι τα πράγματα αρκετά περιπλεγμένα σαν αυτή τη ψηφοφορία. Και θα ψηφίσουμε σε πολλά σημεία ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. Γιατί σε κάθε σημείο θα γύρει η πλάστιγκα προς άλλη πλευρά. Υπαριθμόν 1. Το πολύ υπαριθμόν 1 της έκθεσης γύρω και πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 42. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά για το 42. Βότο 40. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. ανέφερε, Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτεται. Από κοινού. Το κολέγιο υπαριθμών 3 και 14. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτονται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε από εκείνο μια ομάδα τροπολογιών από το 43 δηλαδή μέχρι και την 117 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση σε αυτό το πρώτο πακέτο. Ψηφίζουμε. Ένας παραπάνω για το ΑΕΛΚ και ένας παραπάνω για τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ βγάλτε την κάρτα, συνάδελφα. Εντάξει. Πέρας. Η ομάδα των τροπολογιών αυτών εγκρίνεται. Και τώρα πάμε σε μια άλλη ομάδα τροπολογιών. Στην ομάδα παριθμών 2 που ξεκινά από το 44 και φτάνει ή στο 121 συμπεριλαμβανόμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ομάδα τροπολογιών υπαριθμών 2. Και τώρα πάμε στην ψήφιση της τροπολογίας υπαριθμών 50. Υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφορία για την τροπολογία 50 ψήφισαν όλοι πέρας Το Παγιολάνγκη εγκρίθηκε. Και τώρα με το από το 11 που φτάνει στο 88. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Για την ομάδα 11 έως και 88. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Decadono dunque gli emendamenti 67. 66, 67 και τον 6 καταπίπτουν. Ναι. Οπότε προχωρούμε τώρα στο τρίτο των τροπολογιών που ξεκινούν από το 43 και φτάνουν στο 98. Σας προτείνω να κάνουμε κατευθείαν ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται η ομάδα τροπολογιών. Και τώρα. Ομάδα τροπολογιών. Από το 111 μέχρι και το 113. Και όπως φτιάχτηκε η λίστα ψηφοφορίας, η ομάδα τροπολογιών από το 51 μέχρι το 61 αυτόματα εγκρίνεται ε, λόγω του την κρίναμε την ομάδα τροπολογιών υπαριθμών 3. Οπότε πάμε τώρα στο, στο παγίδο 111 έως και 113. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτουν. Και τώρα. Ομάδα τροπολογιών. 115 έως και 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Οι άλλες καταπίπτουν και πάμε στο 120. 120. Υπέρ. Κατά. Λειτουργικό έλεγχο για την τροπολογία 120. επαλήθευση ψηφίζουμε. Είναι η τροπολογία Μπέντσεν. Πέρασε. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παραδείγματος 43. Καταπίπτει και πάμε στο 6. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 επαλήθευση ψηφίζουμε Πέρας. Εγκρίνεται. πολύ υπερθυμόν 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από κοινού θα ψηφίσουμε το 65 και το 91. 65 και 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 71 και 106 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 113 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 113 Α, ε, διορθώνει πρόεδρος, πρόκειται περί του 13. aperta. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Και κοντράριο και si Αποχές. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Για το 74. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 79 μέχρι και 81 μαζί. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Από το 82 τώρα μέχρι και το 83 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνονται. Ε, συγγνώμη, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 82 και το 83. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνονται 84 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το 84 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 55. Διορθώνει πρόεδρος. 85. Φαβόρε και κοντρά. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για το 87. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά καλύτερα κάνουμε πάλι λήθευση για το 93. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται όντως. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Από κοινό. Από το 100 μέχρι το 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 17. Ψηφίζω. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνεται. Και από εκείνο 111, 112 και 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. από εκείνο 115, 116, 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 117 υπέρ κατά απορρίπτονται και πάμε στην ομάδα 114 έως το 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 115 υπέρ κατά όχι 125 είναι πρόεδρος 125. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Από κοινού τώρα. Όχι. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 125. Ψηφίζουμε. 125. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Όπως είπαμε. 122 και 123 από κοινού. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 122 και 123 θα κάνουμε υπαλήθευση. Ψηφίζουμε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Και πάμε στο 127. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερος έλεγχος για το 128 ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. 18 λέει ο δικός μου της εφορίας, λέει ο πρόεδρος. Α, ζητήσατε για το 130... Επαλήθευση βεβαίως. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Δέκα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωση. Από κοινού τώρα το 19 και το 26. 19 και 26 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 21 ηλεκτρονικά για το 21 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται καταπίπτει το υπαρθμό 22 πάμε στο 23 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το 23. Πέρας. Απορρίπτονται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Από το 27, το 28 και το 29 αλλά δεν ψηφίζονται. Και πάμε στο 30. Μπέντσεν. Α, όχι. Καταπίπτει το 30, λέει ο Πρόεδρος, και πάμε στο 31. Υπέρ, κατά, αποχές. Ευχαριστώ για τη βοηθειά σας, συνάδελφε, αλλά δεν χρειάζεται. Το 31 εγκρίνεται. 32, υπέρ, κατά, αποχές απολύπτεται. Το 34 δεν πρέπει να ψηφιστεί και πάμε στο 38. Είναι τροπολογία ριβαζή, απευθείας ηλεκτρονικά. 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Παρακαλώ ένας από εσάς να βγάλει την κάρτα. Ένας παραπάνω από το έλκα. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40. Μπένσεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε επαλήθευση για το 41. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Γκέρεκ, Αλλά και στους σκιώδες ηγητές που μαζί σας συνεργάστηκαν. Τέλος η ψηφορία. Τα πράγματα κάπως ε, περιπροβλεγμένα, αλλά ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ένα μικρό διάλειμμα λίγο λεπτών, τόσο ώστε όποιος θέλει να αποχωρήσει. Ταχαίως παρακαλώ. Please I Παρακαλώ, συνάδελφοι. Αποχωρήστε ταχύτατα, παρακαλώ, για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσης διάταξης, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το κάνουν με γοργούς ρυθμούς. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τη γνωμοδότηση της κυρίας Βαμπρέντ με θέμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Vorrei ricordare σας υπενθυμίσω εν συντομία κάποια στοιχεία που τα γνωρίζουν όσοι συνάδελφοι που παρακολουθούν το θέμα. Έχουν υποβληθεί σχεδόν 500 τροπολογίες, άπειρες προτάσεις, πληθώρα τροπολογιών από τους συναδέλφους. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας ε, με βάση το άρθρο 54 συνεργάζεται για το θέμα αυτό με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και ο ρόλος της Επιτροπής ΙΤΡΕ είναι πολύ σημαντικός γιατί είναι συνδεδεμένη η Επιτροπή στη διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά, όπως κάνατε και εσείς προηγουμένως, την ε, εισηγήτρια της ε, νομοδότησης για το αξιόλογο έργο της και για τις ε, τακτικές επαφές που είχε με τους σκιώδεις ηγητές. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για ένα πεντάλεπτο ή λίγο παραπάνω το κρίνει απαραίτητο. Κατόπιν θα ακούσουμε τους και οδησηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Καθλίν, έχεις το λόγο. Thank you very much, uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερος τις ευχαριστίες σας προς τους σκιώδης ηγητές και τους βοηθούς μας γιατί ήταν εξαιρετικά πιεστικό το χρονοδιάγραμμα για την γνωμοδότηση αυτή και τα καταφέραμε ε, με κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και με έναν ε, αξιοπρεπή κατάλογο ψηφοφορίας να προχωρήσουμε. Είχαμε 500 κεντρο απολογίε 536. Δεν με φόβησαν αυτές, αλλά έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να συνεννοηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία και με τις άλλες επιτροπές, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Γιατί θα πρέπει να δούμε το χρηματοδοτικό σκέλος, να δούμε τι αποκλειστικέ αρμοδιότητες και τι επιτροπή ΕΚΟΝ, γιατί έχουμε εμεί αποκλειστικέ αρμοδιότητες για τα δικά μα, αλλά θέλουμε σε τελική ανάλυση η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η θέση του να είναι συνεπή. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσουμε ε, έγκαιρα τις διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες επιτροπές για να διατρανωθεί μια συμπαγή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι Ποιε είναι οι αδρέ πολιτικέ γραμμέ. Δεν πρόκειται να επισέλθω στη λεπτομέρεια τη κάθε τροπολογία, αυτό είναι αδύνατο. Οι αδρέ πάντω πολιτικέ γραμμέ ε, είναι σημαντικέ. Αυτέ θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί όπω σα είπα, έχουμε αποκλειστικέ αρμοδιότητε. Θα πρέπει να τι αξιοποιήσουμε, να εμείνουμε σε αυτέ και να επιδιώξουμε καλέ συμφωνίε, που τα καλά να είναι, είναι ότι είναι δυνατέ. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε υπερκομματικές συμφωνίες ε, για μια συμπαγή πολιτική γραμμή. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, είχαμε εκτενείς συζητήσεις και με τον Αρμόδιο και με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Δεν μας βοήθησαν και πολύ. Αλλά καταλήξαμε τελικά σε μια πολιτική γραμμή στις επιτροπές Ήτρε, Τραν, Budget, Econ. Πολύ χρήσιμο αυτό και δεν διάβασα βέβαια, ομολογώ, δεν διάβαζα ακόμη όλες τις τροπολογίες των Επιτροπών Προπολογισμών και Οικονομικών. 1.300 τροπολογίες υποβλήθηκαν. Δεν είμαι καν βέβαιη ότι θα προλάβω να τις διαβάσω όλες από τις δύο επιτροπές. Τα καλά νέα είναι ότι δεν αμφισβητούνται κάποιες προτάσεις ούτε στη δική μας επιτροπή ούτε στις άλλες. Οπότε θα πρέπει με βάση το άρθρο 8 να εξασφαλίσουμε αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή Προπολογισμών και ΕΚΟΝ και να καταλήξουμε σε σωστή συνεργασία. Είμαι πάντω αισιόδοξη. Εμείς έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για το 5.2, για το άρθρο 5.2. Και αυτό το άρθρο περιέχει τρία στοιχεία. Καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα καλό κατάλογο των κριτηρίων και των τομέων προτεραιότητας που είναι η ενέργεια, οι υποδομές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακό θεματολόγιο, έρευνα και ανάπτυξη. Θέλουμε μια σωστή πολιτική γραμμή, λαμβάνοντα υπόψη αν όχι όλες τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων, τουλάχιστον τις περισσότερες από αυτές. Επίσης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, γιατί καλό είναι να έχουμε προτεραιότητες, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε τι είναι εφικτό με τις επενδύσεις και να κάνουμε τη σωστή οριοθέτηση. Αυτό είναι σημαντικό για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχουμε τις νέες πολιτικές για το κλίμα και για άλλους τομείς που οριοθετούν ουσιαστικά το επενδυτικό σχέδιο. Επίσης, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στη συμφωνία για το earmarking, για την προσημείωση των ποσών. Εγώ πρότεινα ένα μόνο earmarking, γιατί πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση αυτή της ενεργειακής απόδοσης. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες ενισχύοντας αυτή τη θέση και μάλιστα οι περισσότερες πολιτικές ομάδες επιδιώκουν ενίσχυση αυτής της θέσης. Αυτή είναι η δική μου πολιτική γραμμή και υπάρχουν ερωτηματικά για αυτό το θέμα. Ένα άλλο earmarking αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόσες επιδοτήσεις ε, ε, από την ΕΤΕΠ και από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε στη συζήτηση σήμερα να συνδυάσουμε αυτά τα δύο θέματα, γιατί περισσότεροι θέλουν να δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που αναγνωρίζουμε και εμείς, αλλά αλλά να μην δώσουμε επιταγή λευκό στην ΕΤΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χαράξουμε τις γραμμές μας και να, δούμε, να πούμε που θέλουμε να κατευθυνθούν οι επενδύσεις γενικώ. Επίσης για τη διακυβέρνηση. με τροπολογίες μου προτείνω τις κατεξιδότηση πράξης, όπως και οι Επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικών. Η συμφωνία όμως μεταξύ της ΕΤΕΠ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αφορά τεχνικά μόνο θέματα και όχι το περιεχόμενο, την ουσία. Και αυτό το διατρανώνω. Το περιεχόμενο θα πρέπει να αναφέρεται στον κανονισμό που λέει που θα πρέπει να κατευθύνονται σε τι να προορίζονται οι επενδύσεις. Είχαμε ήδη δύο τεχνικές συναντήσεις με τους βοηθούς ε, και τους υπαλλήλου. Ήδη εκπονούμε τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και θέλουμε παρακαλώ τους συναδέλφους να ανασκουμποθούμε αυτή την εβδομάδα για να ολοκληρώσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες Έχω χρόνο και την επόμενη εβδομάδα, αλλά δύσκολα θα είναι την επόμενη εβδομάδα, γιατί ένα τίμα είναι γαλάζια και μετά η επόμενη γαλάζια και μετά έχουμε την ψηφοφορία, οπότε καλό θα ήταν να εντατικοποιήσουμε τις εργασίες αυτή τη εβδομάδα για να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες και να είμαστε διαλλακτικοί, να αφήσουμε τις λεπτομέρειες, να επικεντρωθούμε στις αδρές πολιτικές γραμμές. Ευχαριστώ Καθλή. Οπότε έχει ήδη γίνει σημαντική προεργασία, αλλά έχουμε και πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Προχωράμε τώρα με τους σκιώδης ηγητές. Ο κύριος Έλερ, που είναι ο σκιώδης ηγητής από το ΕΛΚ, έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Να θέσω πέντε σημεία, αλλά πριν από αυτό να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι είναι αγωνίστρια. Να την ε, διαβεβαιώσω ότι είτε πάρουμε τα χρήματα αυτά ε, Τώρα είναι η στιγμή να πολεμήσουμε. Ό,τι, θα κάνετε, ό,τι λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι θα σας υποστηρίξει η ομάδα μας σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Συμφωνεί το ΕΛΚ να, δι... να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του ετήσιου προπολογισμού και η μοναδική διαφορά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν θέλουμε να προδιαγράψουμε θέματα ε, χρηματοδότησης για τον ορίζοντα 2020. Θέλουμε να εξαιρέσουμε την δυνατότητα να υπάρχει εξαίρεση επειδή υπάρχει καλή επίδοση και οι αρχές χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να κοιτάξουν μόνο το ένα αλφα. Έχουν ήδη ζητήσει ευελιξία σε ό,τι αφορά το συνέδριο του προπολογισμού και νομίζουμε ότι θα πρέπει να βρούμε μία λύση όπως έχει βρεθεί στο παρελθόν. Πιο πολλά χρήματα για καινοτομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ΕΛΚ μαζί με τις άλλες ομάδες ζητά πιο πολλά χρήματα τα, για δραστηριότητα για δραστηριότητε που ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Στρατηγικών Επενδύσεων σε ό,τι αφορά και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θέλουμε 3 δισεκατομμύρια επιπλέον να πάνε σε, στα πλαίσια του IEF. Υπάρχει τεράστια μόχλευση σε ό,τι αφορά τα ποσά αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μέχρι και 1,28 αυτό ήταν βασικό λοιπόν ζήτημα στη θέμα της γενικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Άρα τα εφιστάμενα εργαλεία υπάρχουν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν έλλειψη σε επενδύσεις κινδύνου. Αυτό δεν είναι μυστικό. Και για την δημιουργική βιομηχανία θα θέλαμε να το το θέμα αυτό ότι η δημιουργική βιομηχανία και το ICT είναι σημαντική προτεραιότητα. Αυτό νομίζω ότι βρίσκει σε πολλέ ομάδε, βασική πολιτική και δεν πρόκειται για εξυπηρέτηση μόνο ενό κλάδου. Απασχολεί πολύ όλη την Επιτροπή. Να μην υπάρχει πολιτικοποίηση τη διακυβέρνηση του, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΤΣΙ. Η ανάληψη υψηλού κινδύνου στις επενδύσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία εξέτασης και θα πρέπει να κοιτάμε τι έργα χρηματοδοτούνται και για ποιους τομείς χρηματοδοτούμε, Θα πρέπει να μην έχουμε ένα ευχολόγιο εδώ στον κανονισμό, να βρούμε συγκεκριμένους τομείς προτεραιοτήτων Κριτήρια επιλεξιμότητας επίσης, ή δεν πρόκειται να πετύχουμε αν μπούμε σε υπερβολικό βαθμό λεπτομέρειας, θα χάσουμε. Και εδώ θα υπάρχει και κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Τελευταίο θέμα. Πράξει κατά εξουσιοδότηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πράξει κατά εξουσιοδότηση για τη συμφωνία έτσι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για το μέλλον, για τι καταστηντηρίες γραμμέ επενδύσεων που θα καταρτιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. όχι υπερβολικές λεπτομέρειες, αλλά δύο πράξεις κατά αξιοσυνδότηση για την ε, κατασκευή και για τις κατευθυντηρίες γραμμές. Γιατί άλλα θα χάσουμε στον αγώνα αυτό. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Τουσενόφσκι από τους ε, μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Βαμπρέντ γιατί το πιστικό χρονοδιάγραμμα ε, ε, δεν ε, είναι ευνοϊκό και βολικό για τέτοια πληθώρα τροπολογιών. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να διασπαστεί η προσοχή μας, γιατί είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη, στις αδρές γραμμές. Καταρχήν, από πού θα βρεθούν τα κονδύλια. Πιστεύω ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι στα άρθρα 18 και 19. Επίσης πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να πάρουμε λεφτά από το ορίζοντας 2020 και το συνδέοντας στην Ευρώπη, το μηχανισμό αυτό, γιατί έτσι θα περιπλέξουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι από πού θα βρεθούν τα κονδύλια. Η ομάδα μου είναι κατά οποιοδήποτε ανοίγματο συζητήσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το έχουμε ήδη πει και θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να παρέμβουμε σε θέματα της πολιτικής συνοχής. Γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. και ίσως ε, υπονομεύσουμε τις μέχρι τώρα συμφωνίες. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις αποκλειστικές μας αρμοδιότητες και να μην χάσουμε την ευκαιρία να επενδύσουμε στις ψηφιακές υποδομές και στην ενέργεια, όπως είπε και η συγγήτρια. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ταυτόχρονα δεν συμφωνώ με το υπερβολικό ευχολόγιο. Θα πρέπει να μείνουμε σε γενικό επίπεδο και να μην προσθέτει ο καθένα τις δικέ του προτεραιότητε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ενδιαφέροντα προγράμματα και σχέδια. Δεν συμφωνώ με το earmarking, με τον ειδικό προορισμό κάποιων κονδυλίων. Είμαι κατά του ειδικού προορισμού των κονδυλίων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο. Και φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις μεσαίες κεφαλαιοποίησης στα κονδύλια αυτά. Και να έχουμε και ένα ελάχιστο αριθμό κριτηρίων επιλεξιμότητας. Είμαι υπέρ μια καθαρής δομής, μιας ε, συγκροτημένης δομής, όπως είπε και ο κύριος Έλερ, που υπέβαλε πολύ λογική πρόταση. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και είμαι, στα, στο, στη διάθεσή της και θα σταθώ στο πλευρό της, γιατί επαναλαμβάνω πιεστικότατο το χρονοδιάγραμμα και τεράστιος φόρτος εργασίας, λόγω και της πληθώρας των τροπολογιών. Ο κύριος Φέντερλε τώρα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον κύριο Τεμπάκερ που είναι ο σκιώδης ηγητής ε, και ζητά συγγνώμη για την απουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για το έργο που επιτέλεσε με του βοηθού και το επιτελείο τη, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο αριθμό των ανθρωπολογιών που θα πρέπει να εξετάσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πιεστικό το χρονοδιάγραμμα, εξαιρετικά σημαντικό το θέμα και παραλαμβάνω καταιγισμό τροπολογιών. Είχαμε ήδη αρκετέ συναντήσει με του κέρδη ηγητέ, ε, τα πράγματα ακολουθούν το σωστό δρόμο. Δεν θα σταθώ σε λεπτομέρειε, ε, όπω και οι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνω τι ε, βασικέ γραμμέ των φιλελευθέρων. Ξεκινώ με ένα θέμα που είναι κοινό μα μέλημα. Από πού θα προέλθουν τα κονδύλια συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να προκύψει ούτε από το ορίζοντας 2020 ούτε από το μηχανισμό συνδέοντας, Ευρώπη, την Ευρώπη. Και μάλιστα ακόμα και το ελεκτικό συνέδριο θα βάλει για το κατά πόσο είναι καλή αυτή η ιδέα. Και είναι και πολιτικό το μήνυμα. Θα πρέπει να βρεθούν από αλλού τα κονδύλια και έχουμε πολλέ ευκαιρίε στον κοινοτικό προπολογισμό. Αναξιοποιεί κονδύλια, περιθώρια ή το, το μηχανισμό ελαστικότητα. Επίση, ε, ε πού θα, θα θέλαμε να ξοδέψουμε αυτά τα χρήματα. Τι θα χρηματοδοτήσουν οι επενδύσεις. Θα συστήσουμε ένα επενδυτικό ταμείο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που θέλουμε να προσελκύσει ειδικό, ιδιωτικό κεφάλαιο και θα τους υποδείξουμε που θα ξοδέψουν τα χρήματα. Για να είναι λειτουργικό το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και να προσελκύει ιδιωτικά κονδύλια, θα πρέπει να είναι σχετικά ελαστικό. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρό ο προπολογισμό με συγκεκριμένε οδηγίε. Επίση, συμφωνώ να έχουμε κάποια κριτήρια, αλλά δεν συμφωνώ να αρχίζουμε να προβλέπουμε κονδύλια ειδικού σκοπού και να υπαγορεύουμε στου επενδυτέ που θα πρέπει να επενδύσουν. Αν έχουμε ένα ενδιαφέρον επενδυτικό πρόγραμμα, είτε στι μεταφορέ, στην ενέργεια ή στο ψηφιακό τομέα, να μπορούν να έχουν ελεύθερη επιλογή οι επενδυτέ. Επίση, το θέμα τη διακυβέρνηση. Ε, θα πρέπει να αφήσουμε την ε, Επιδετική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο μακριά από πολιτική επιρροή. Δεν θέλουμε πολιτικοποίηση του Ταμείου. Να βρίσκουν αυτά τα αρμόδια όργανα με βάση αξιοκρατικά κριτήρια τα σωστά επενδυτικά προγράμματα. Επίσης να βρούμε τη σωστή ισορροπία για την ανάμειξη των ε, κρατών μελών και των εθνικών τραπεζών πρόθεσης. Δεν μιλούμε εδώ για συζήτηση πολιτικών και ε, ομάδων ή κομματικών συζητήσεων. Ε, προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την κρίση, να κινητοποιήσουμε κεφάλαιο για να εξασφαλιστεί και πάλι απρόσκοπτη επενδυτική ε, ροή, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε τρύπε στον προπολογισμό. Θέλουμε ένα λειτουργικό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων, γι' αυτό είμαστε καλά των κονδυλίων ειδικού σκοπού και κατά της υπερβολικά άκαμπτης διακυβέρνησης. Ο κύριος Κλωτ Τουρμές από τους Πράσινους, παρακαλώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Κατλέν και τους ε, συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς προσπάθησαν να ενσωματώσουν τις τροπολογίες σε συμβασμούς ως πράσινοι. Ένα από τα βασικά μας μελήματα είναι να προστατεύσουμε τον προπολογισμό για την έρευνα. Νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μεγάλο λάθος ε, καταστρέφοντας ε, ένα από τα σημαντικά, μια από τις πιο σημαντικές γραμμές ε, του προπολογισμού για την έρευνα και σύμφωνο που υπάρχει ευρία ομοφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Άλλη ανησυχία που έχουμε, η τεχνική αρρωγή. Και ποια είναι η πραγματικότητά της κοιτάω ότι πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην τελική ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει πολύ για την ε, ανάγκη επιπρόσθετης τεχνικής αρρωγής, αλλά κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία, μόνο 20 εκατομμύρια προσθέτουν στην υφιστάμενη τεχνική αρρωγή. Κάποια προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει στο παρελθόν με 20 εκατομμύρια τεχνικής αρρωγής από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε μία ομάδα 10-15 ατόμων. Αυτό, τελεία και παύλα. Άρα έχουμε έργα με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τάξεως των 10-15 εκατομμυρίων και αυτό δημιούργησε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέσεις για 10-15 άτομα. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της θεωρίας αυτών που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της πραγματικότητας. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τα χρήματα αυτά στη τελική ανάλυση θα κατευθυνθούν στο τομείς που έχουμε δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση του ECR και των φιλελευθέρων να είμαστε κατά του ειδικού προορισμού, του earmarking. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται earmarking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ή άλλως, δεν θα υπάρχει επαρκή τεχνική αρρωγή και τελικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πάρουν τα χρήματα τα οποία ελπίζουμε να πάρουν. Και ο άλλος τομέας όπου ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και από προηγούμενα προγράμματα είναι σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας έχουμε ένα κενό, ένα χάσμα 50-60 εκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις και η Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων τα έχουν εντοπίσει αυτά. Ξέρουμε ότι τα κονδύλια που δημιουργήσαμε, τα ταμεία που χρησιμοποίησαμε πριν από 4-5 χρόνια, ένα παράδειγμα ενό ταμείου το οποίο διαχειρίζεται η Deutsche Bank. Συνεπάγονταν ε, δισεκατομμύρια επενδύσεων. Μιλάμε δηλαδή για παράγοντα μόκλευσης 15, 15 πλάσιο και σε θέματα ελληνικής αποδοτικότητας. Και θέλουμε δύο λοιπόν earmarking για τις μικρομεσαίες και για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο θα έδινε μεγάλη όθηση στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, μια στιγμή που υπάρχει απελευθέρωση ουσιαστικά των τιμών ενέργεια και αύξηση τους ασφαλώς. Ένα τελευταίο ζήτημα για τη διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρούμε τα βασικά κριτήρια για το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα και θα πρέπει να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή. Για να δούμε λοιπόν τι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί αν δεν το πράξουμε αυτό, ουσιαστικά δεν είναι λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η συμφωνία με την Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Από την ΚΟΕ η κυρία Ένστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εξ ονόματο τη συναδέλφου Παλώμα Λόπε, η οποία δεν μπόρεσε να πραγματευτεί σήμερα εδώ. Θα ήθελα και εγώ καταρχά να ευχαριστήσω του σκιώτε, όπω και την εισηγήτρια ασφαλώ, για την όλη διαδικασία και την ε, ταχύτητα. Αυτό αφενό. Ξέρετε ότι είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί και είμαστε επικριτικοί εξ αρχή ε, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Απαράδεκτο το γεγονός ότι οι δημόσιες εγγυήσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να γίνουν σε μια χρονική συγκυρία όπου υπάρχουν υποσχέσεις για δημόσιες επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα και στην οικοδομία. Αυτό το παραμελούμε ολοκληρωτικά. αυξάνεται το κόστος για του φορολογούμενου. και αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα σε θέματα που μα δυσκολεύουν ιδιαίτερω. Το θέμα αυτό λοιπόν θα το θέσουμε και αύριο σε θέματα τέτοια προβληματική. Να μπω πιο συγκεκριμένα σε κάποιε λεπτομέρειε. Είναι δύσκολη για μα η απόφαση και η επιλογή των έργων. Δεν συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Πολύ δύσκολο αυτό ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει. Η απόφαση λοιπόν για το πώς θα επιλεχθούν τα προγράμματα, ποια θα επιλεχθούν, όλα αυτά είναι πολύ αναπαρκώς ρυθμισμένα. Επόμενο σημείο. Όπως και, εμείς, όπως και οι πράσινοι εμείς πιστεύουμε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να συνδέεται με το στόχο, με τη στόχοθέτηση. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την αγορά ενέργειας θα πρέπει να υπάρξουν οικονομίες. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάγκης επενδύσεων σε διάφορα κράτη-μέλη. Επόμενο σημείο, κοιτώντας τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ιδιαίτερα η περιφερειακή και τοπική συνοχή πρέπει να προωθεί Άρα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να προωθηθούν έργα για κατασκευές, για αυτοκινητοδρόμους, όχι. Χρειάζεται και κοινωνικά project. Ένα τρίτο των ε, μέσων των κονδυλίων θα πρέπει να είναι προορισμένα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται και από τις ε, τροπολογίες μας. Άρα, συνολικά θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί παιχνίδι βουντού. Όπου το μόνιμο ερώτημα είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Ορίζοντα 2020 και ένας τέτοιος ε, αντίκτυπος μόχλευσης δεν θα υπάρξει σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που αφαιρούνται από τον ορίζοντα 2020 και δεν βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση αν υπάρξουν θετικέ επενδύσει πιο καλά από ό,τι στον δημόσιο κλάδο. Άρα συνολικά πολύ επικριτικοί είμαστε για το θέμα αυτό και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να σημειώσουμε μια οικονομική πρόοδο, μια οικονομική εξέλιξη σωστή. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των αγορτών από τους και δυσυγητές και τώρα πάμε στα υπόλοιπα της Επιτροπής. Παρακαλώ, συμμορφωθείτε πάντως και με τα χρονικά όρια. Πρώτη πρώτη η κυρία Πιλάρ το λόγο Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω τον ερμό των ε, προελισάντων. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όχι μόνο για το κολοσσιαίο έργο που επιτέλεσε, αλλά και για την πολύ σαφή και περιεκτική παρέμβασή της ε, προηγουμένως, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι τα ουσιώδη σημεία. Τώρα, πού θα δαπανίσουμε τα κονδύλια. Ο κύριος Έλερ παρουσίασε τη γνώμη τη θέση του ΕΛΚ. Είναι σαφής. Κάτω τα χέρια από το ορίζοντα 2020 και από το συνδέοντα στην Ευρώπη να βρεθούν από τον γενικό προπολογισμό ίσως. Τώρα, αυτό για την προέλευση των κονδύλιων. Τώρα για τον προορισμό τους, που είναι και αυτό θέμα που ενδιαφέρει την Επιτροπή Ήτρε, μπορούμε να συζητήσουμε πόσα κονδύλια ειδικού σκοπού, ειδικού προορισμού θα έχουμε πόσα markings Μπορούμε να έχουμε γενικά κονδύλια ειδικού σκοπού, πιο εξατομικευμένα, πολύ πιο εξειδικευμένα. Θα το δούμε. Θα μπορούσαμε ίσως, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα της Ήτρε, να προβλέψουμε κάποιους δείκτες, να δώσουμε κάποιες ενδείξεις ότι μας ενδιαφέρουν η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης να τονίσουμε να το, τη σημασία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 που αφορά τις διασυνδέσεις για την ηλεκτρική ενέργεια. Την είναι σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φάνηκε και από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου και από το Συμβούλιο Κορυφής προηγούμενης εβδομάδας. Επίσης, θα πρέπει γενικά να λάβουμε υπόψη ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, τη χρήση των ε, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Γιατί και στον τομέα της ενέργειας οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας συμβάλλουν τα μάλα και συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Έτσι γίνονται και οι απαραίτητες οικονομίες στην ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στις τροπολογίες μας. Γιατί καλό θα ήταν αν έχουμε earmarkings να έχουμε κάποιο ε, γενικό πλαίσιο για τα κονδύλια ειδικού σκοπού και να προσθέσουμε κάποιες ενδείξεις για το πόσο θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν. Ευχαριστώ Πιλάρ, κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω και τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια προς την Κάθλη για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα και για αυτό που της έχει απομείνει. Σίγουρα δεν είναι λίγο πράγμα. Έχει 1.300 τροπολογίες μόνο από την Επιτροπή Προπολογισμό να εξετάσει. Όλοι είπαμε ε, ότι χαιρετίζουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητά του, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός το ΕΦΣΥ το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι μέσο για την υλοποίηση του σκοπού μας. Ένα τμήμα του ε, προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται αποτελεσματικά είναι το ορίζον 2020. Και το γεγονός ότι υπάρχει υπερκομματική συνένεση και ε, συμφωνία όλων των επιτροπών να διαφυλάξουμε τον προϋπολογισμό του ορίζοντος 2020 γιατί είναι από τα κομμάτια του προϋπολογισμού τα αποτελεσματικά είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η υπερκομματική συνένεση λέει πολλά και θα ήταν είναι μεγάλο λάθος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν δείχνει ελαστικότητα αυτή τη στιγμή είτε προς επιτροπές είτε προς τις πολιτικές ομάδες. Μέχρι στιγμής φαίνεται αδιάλακτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει και εμείς ε, να σταθούμε αμετακίνητοι εμένοντας ε, πιστά στην προάσπιση του ορίζοντας 2020. Επίσης, ε, σημασία της διακυβέρνησης. Γιατί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις υποδομές. Σημαντικές βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το μέλλον και με σωστές δομές διακυβέρνησης θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές επενδύσεις μέσω του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων φτιάχνοντας την οικονομία του μέλλοντος είτε μέσω του πολιτισμού, είτε μέσω των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, είτε της τεχνολογίας και ανάπτυξης και της έρευνας. Αλλά σίγουρα η διακυβέρνηση είναι θεμελιώδες συστατικό και θα πρέπει να βρει τη θέση της στον, στον κανονισμό, συγγνώμη, όπως άλλωστε προ... προανήγγειλε και η Κάθλιν. Η κυρία Τελίτσκα από τους Ο κύριος Τελίσκα, συγγνώμη, από του Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφο Φρέντερικ ε, Φέντερλε. είμαι λοιπόν σύντομο. Καταρχά, εκτιμώ το έργο της συγγήτριας. Πολύ απαιτητικό. Εκτιμώ ιδιαίτερα και τον ανοιχτό χαρακτήρα τον οποίο επιδεικνύει σε ό,τι αφορά τα σχόλια των άλλων συναδέλφων από τι άλλε πολιτικέ ομάδες. Να τονίσω ένα σημαντικό στοιχείο. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων εδώ και καιρό αποτελεί το πιο σημαντικό project τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο ω χρηματοοικονομικό μέσο, αλλά ω πολιτικό έργο. Αν αποτύχουμε αυτή τη φορά, θα υπάρχει σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει Εμεί, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να το κάνουμε και να το δημορφώσουμε σωστά. Για να το δημορφώσουμε σωστά θα πρέπει να έχουμε και να δημιουργήσουμε επαρκή εμπιστοσύνη στους ιδιωτικούς κυρίως επενδυτές. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τονίσω αυτό που ήδη έχει αναφερθεί, ότι θα πρέπει από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει η λιγότερη δυνατή πολιτική παρέμβαση. Γιατί αν τα παρακάνουμε, θα χάσουν την εμπιστοσύνη του οι ιδιωτικοί επενδυτέ. Και εξαρτώμαστε από αυτού. Άρα, ω εκ τούτου, πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για του επενδυτέ. Γι' αυτό λοιπόν να υπογραμμίσω κάτι το οποίο φαίνεται να παραμελούμε στι δηλώσει μα. Πρόκειται για έναν από του τρει πυλώνε του σχεδίου Juncker. Η Άλλο δύο πυλώνες είναι εξίσου σημαντικοί, ίσως και πιο σημαντικοί. Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να μην υπάρξει earmarking, ειδική ανάθεση με ποσοστιαίες ε, τέτοιες, με ποσοστιαίους ε, τουρισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια διατύπωση για να τονίσουμε ότι αυτή την έμφαση δίνουμε, αυτή την επένδυση θέλουμε να κάνουμε στους ταχαίους αυτούς αναπτυσσόμενους ε, κλάδους, αλλά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να ορίζουμε ποσοστά, θα υπάρξει μια πολιτική άσκηση για την πραγματευσή τους. Τέλος, από πού θα πρέπει να προέλθουν τα χρήματα για τις εγγύησεις. Να ενισχύσω την ομοφωνία, τη συνένεση που υπάρχει, ούτε ορίζοντας ε, 2020 του συνδέοντα στην Ευρώπη. Για τον εξή λόγο, ότι το συνδέεται στην Ευρώπη προορίζεται για πολύ διαφορετικά έργα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ενωμετικό Ταμείο, Γιατί ευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία συνήθω δεν έχουν απόδοση στην επένδυση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εμπρογνωμοσύνη τη προτείνει κάτι το οποίο δεν έχει καμία λογική. Αφήστε που έχει δημιουργηθεί εν μέρη το συνδέεται στην Ευρώπη από την χρηματοδότηση για τη σύνοχη. Αυτό θα δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα, επιπλέον αντίσταση από κάποιε χώρες. Σα υποστηρίζω λοιπόν, αλλά σα παρακαλώ πάρτε υπόψη και τα σχόλιά μας. Καλή τύχη και ελπίζω να καταφέρετε να φέρετε σε ίσο τέλος την ε, θέμα αυτά. Η κυρία Πινιέρα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο και τη διαβεβαιώ για την αμέριστη συνεργασία μας και το μελλοντικό της έργο. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τον προϋπολογισμό του ορίζοντα 2020 και επίσης να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό να φανεί αυτή η υπερκομματική συμφωνία, αυτή η ενότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ της διαφύλαξης του προϋπολογισμού του ορίζοντας 2020. Εν θα πρέπει να φανεί αυτή, αυτό το πνεύμα ενότητας και σύμπνοιας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ε, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές κατέθεσα τροπολογίες που αναφέρονται αφενός στη διακυβέρνηση και αφετέρου στις ε, επιδιώξεις μας. Ε, δηλαδή όχι μόνο για το τι είδος ε, επενδυτικά σχέδια θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά και ε, τι επιχειρήσεις. Επιμένουμε στη διαφάνεια, θα πρέπει να εφαρμόζονται διαφανή κριτήρια, να υπάρχει λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα κριτήρια και τους λόγους απόρριψης κάποιων σχεδίων. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε όχι μόνο τι είδους δραστηριότητες και σχέδια θα γίνουν, αλλά και τι είδους επιχειρήσεις θα αναλάβουν αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις αρχές και τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε επιχειρήσεις ε, που είναι υπέρ της ισότητας των φύλων ε, ε, και των μισθών και να μην κάνουμε αξιολόγηση, να μην επαληθεύουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις με κονδύλια κοινοτικά γίνονται προς επιχειρήσεις που όντως εφαρμόζουν τα κριτήρια της ισότητας των δύο φύλων, των ίσων, μισθών για ίση εργασία και της ε, εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Αλλά κολέγα, Κύριε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ασφαλώ να συγχαρώ την Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το έργο της. Εν και των διακοπών του Πάσχα. Να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος Έλερ για τη διακυβέρνηση. Και ξέρω ότι υπάρχουν διάφοροι που προτείνουν η διαχείριση, η διακυβέρνηση να συμπεριλαμβάνει και την εποπτεία τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω στου συναδέλφου ότι αυτό που συζητάμε, το Ταμείο Επενδύσεων, είναι ένα Ταμείο Εγγύσεων 8 ε, δισεκατομμυρίων. Ελπίζουμε να προσελκύσει 300 δισεκατομμύρια ιδιωτικού πόρου. Οι ιδιωτικοί επενδυτέ λοιπόν, φαντάζεστε, να βάζουν λεφτά κάπου που θα αποφασίζουν οι πολιτικοί. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι αυτό και δυστυχώ δεν έχουμε καλή φήμη δεν έχουμε την καλύτερη φήμη για να είμαστε καλοί επιχειρηματίες. Εμείς ε, τι σκοπό, τι, τι καθήκον έχουμε να θέσουμε τους κανόνες και να αφήσουμε το παιχνίδι να ξεκινήσει. Πολιτική συμμετοχή στις κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι να ορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλά μετά το παιχνίδι θα πρέπει να εξελιχθεί από μόνο του. Να θυμάστε ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε δυτικού πόρου. Αν δεν προσελκύσουμε δυτικού πόρου, δεν θα έχει καθόλου νόημα αυτό το, αυτή, αυτό το εγχείρημα. Και αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Ευχαριστώ. Κυρία Μουράνο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και από μένα, Καθηλήν περιμένουμε πολλά από την γραμματότησή της και τη στήριξη των θεών μας. Γνωρίζουμε ότι αυτή, μα αυτό το οσανά εξ ουρανού από το επενδυτικό, από Στρατηγικών Επενδύσεων ε, το περιμένουν πώς και πώς ε, οι επιχειρήσεις και οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τη δυνατότητα και στους περιφερειακούς φορείς και τις τοπικές αρχές που έχουν προϋπολογισμό να συμβάλλουν ε, στην δρομολόγηση των επενδυτικών ε, σχεδίων. Γιατί πολλές, πολλοί οργανισμοί περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην ε, Γαλλία έχουν προϋπολογισμό και είναι κρίμα να μην συμμετέχουν σε επενδυτικά σχέδια, χάνοντας έτσι δυνατότητα να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών ε, ε, Επενδύσεων εφόσον το επιθυμούν. Θα ήθελα να ανοίξουμε και στις, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το ταμείο. Οπότε στο άρθρο 19 θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορούν και οι περιφερειακοί τομείς να στηρίζουν επενδυτικά σχέδια. Να μην κλείνουμε καμία πόρτα, αντίθετα να ανοίγουμε πόρτες εκεί που μπορεί να βρεθεί συμπληρωματική χρηματοδοτική στήριξη για την ε, χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Έχω ε, κατά νου μία δύσκολα χρηματοδοτωμένη υποδομή που είναι όμως απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Γαλλίας που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Να ανοίξουμε λοιπόν το ταμείο αυτό και στις περιφερειακές αρχές ε, για να ενισχύσουμε και την αποκέντρωση, ιδιαίτερα σε κράτη που επιτρέπουν τέτοια δυνατότητα. Συνάδελφος Γκρίφιν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και πάλι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καθλίν για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει, αλλά και για την πολιτική ηγεσία που έχει επιδείξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια προσέγγιση από τα μέλη όλων των ομάδων εδώ και στην Επιτροπή μας αλλά και στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση του ορίζοντα 2020 και του συνδέοντα στην Ευρώπη. Να δούμε λοιπόν στο θέμα του πού πηγαίνουν τα χρήματα, γιατί προορίζονται τα χρήματα. Βλέπουμε ότι τα καινοτόμα τοπικά έργα που δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην τοπική ανάπτυξη και οδηγούν σε ποιοτικέ βιώσιμες θέσει εργασία μπορούν να υποστηριχθούν από το έτσι. Επίση, ε, μιλήσατε, Κατλέιν, για την ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. και θα πρέπει να, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα πρέπει να επενδύουμε σε τομεί ανάπτυξη όπως η δημιουργική βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Τερέζα. Ο κύριος Έλερ να δευτερολογήσει. Έχουμε λίγο χρόνο. για να διευκρινίσω τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Καταρχά, αν αποτύχουμε και δεν είμαστε ενωμένοι στο θέμα του προπολογισμού, θα χάσουμε. Αυτό είναι ο παράγοντα μόχλευση που έχουμε. Κατά δεύτερον, το θέμα του earmarking και των προτιμήσεων. Θα πρέπει εδώ να βρούμε ένα συμβιβασμό. Η θέση τη ΣΥΤΡΕ δεν είναι τόσο ισχυρή για το θέμα αυτό. Εδώ μπορεί να υπάρχει πιο έντονη διαμόρφωση τη θέση τη ΙΚΟ και τη ΜΠΑΤΖ. Να δώσουμε κάποια αλφα έμφαση. Αυτό, αν το πετύχουμε, μπορεί να δουλέψει. Αν ε, επέμβουμε πολύ και παρέμβουμε πολύ στα νερά των αλληλοπιτροπών, μπορεί να μην πετύχουμε τίποτε. Αυτό που θα μπορούσαμε να αντιπραγματευτούμε στην πραγματικότητα είναι οι πράξει κατά αξιοδότηση. Αν υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τι πράξει κατά εξουσιοδότηση, θα είναι με μια πάρα πολύ ισχυρή θέση ω εισηγητή ένα ανεπίσημο, μια ανεπίσημη συμφωνία για το πώ θα διαμορφωθεί ε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Πολύ πιο πολύ από τις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στην Επιτροπή μα. Γιατί αυτό το πετυχαίνουμε συνήθως με την πρώτερη επεξεργασία και του τους συμβιβασμού για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Αν υπάρχουν ήδη προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Αν θέλουμε λοιπόν κάτι να πετύχουμε, κάτι απτό, το σημαντικό είναι να ζητήσουμε τις δύο πράξεις κατεξουσιοδότηση για το πώς θα τα κονδύλια. Οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν στο μέλλον. Και τώρα το πώς θα λειτουργήσει η δομή της διαχείρισης της διακυβέρνησης. Και έτσι θα έχουμε κάτι απτό. Αν έχουμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, ως εισηγήτρια θα έχετε κάποιο πολιτικό βάρος για να κάνετε κάποιες πρώτες, πρώτερες και να ξέρουμε μία ιδέα για το τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτά. Εξαγάγω συμπέρασμα από τις ισορροπίες εδώ στην Ήτρε. Συμβιβασμό για τις προτεραιότητες, αλλά σε καμία περίπτωση να μην αποδυναμώσουμε τις απόψεις μας με ένα ευχολόγιο. Αλλά να είμαστε σταθεροί και μετακίνητοι για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, για το τι θα αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει άλλη πράξη κατά εξουσιοδότηση, θα παραμείνουμε πάντα στο το παιχνίδι. Ιδάλλω πιστεύω ότι θα αποδυναμώσουμε την άποψή μας, θα αποδυναμώσουμε τη θέση μας, φορτώνοντας υπερβολικά αυτά που επιθυμούμε. Έχει ζητήσει να ευθρολογήσει ξανά ο κύριος Τούρμες. Και εγώ έχω κάνει τέτοιες διαπραγματεύσεις για μια σειρά οδηγιών θα πρέπει να είναι σαφή και αν θέλουμε να είναι προτεραιότητα η πολυμορφή τη ενέργεια και η τότε θα πρέπει κανεί να έχει σαν αφετηρία κάτι που έχει ε, κάποια ουσία, όπω ε, τέτοιο γερμαργή. Αλλιώ δεν θα έχουμε κανένα είδου πυγμή στι διαπραγματεύσει. Άρα αυτά λέει η δική μου ανάλυση, γιατί έχω κάποια πείρα από διαπραγματεύσει. Grazie. Πρόεδρος. Έχουμε πολλές προτάσεις για την Καθλήν. Και τώρα θα δώσουμε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα να σχολιάσω έξι σημεία. Δεν θα σε εκπλήξω αν το πρώτο εξ αυτών είναι ο προπολογισμό. Να σας πω γιατί μας προβλημάτισαν αυτά τα οποία ακούσαμε στην Επιτροπή σας και σε άλλες επιτροπές να απαλείψουμε το 18 και το 19. Να σας εξηγήσω ακριβώς γιατί μας έχει ανησυχήσει αυτό που ακούσαμε, γιατί από νομικής πλευράς δεν είναι δυνατόν το ΕΦΣΙ να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη χρηματοδότηση. Ξέρετε τι προβλέπει η συνθήκη, ότι η πρόταση θα πρέπει να συνάδει με το πλαίσιο αυτό το, το πολιετές πλαίσιο. Αλλιώς, εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση τέτοια, 8 εκατομμυρίων ας πούμε, δεν είναι νόμιμη συγκρότηση. Επίσης, είπαμε για κάποιο είδους ε, ετήσια ε, συζήτηση και αυτό μας προβληματίζει. Ό,τι δηλαδή, και δεν το χειρότερο αυτό, ότι θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο χάος από το υπάρχουν τώρα. Αλλά αυτό μας ενισχύει ακόμη περισσότερο και έτσι δεν θα προβάλλεται αρκετά η δυνατότητά μας να προγραμματίζουμε τις δαπάνες. Γιατί έχουμε ένα σωρό ε, κρεμούντα ποσά ε, τα οποία θα πρέπει να εκταμιευθούν μέχρι το 2020, τη μία χρονιά μετά την άλλη. Αλλά δεν θα ξέρουμε, αν γίνει έτσι, πόσα θα είναι διαθέσιμα για το κάθε πρόγραμμα. Κατά τρίτον, υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος υποβάθμισης. Και δεν μιλώ για υποβάθμιση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μιλώ για την υποβάθμιση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχουμε 26 δις πληρωμές που δεν έχουν καταβληθεί. Και αν έχουμε άλλες 16 δισεκατομμύρια εγγύσεις για αυτή την υπηρεσία τότε κινδυνεύουμε να υποβαθμιστούμε. Ξέρετε ότι οι Standard Poor's ήδη υποβάθμισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε άμα γίνει κι άλλη ε, υποβάθμιση τότε δεν θα είμαστε επιλέξιμοι για μια σειρά επενδυτών. Επίσης η προσθήκη του 1α ως ε, κεφαλίδας είναι ε, λογικό. Τώρα το κεφάλαιο 1β δεν μπορεί να γίνει, να αλλάξουμε τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις και όπως ξέρετε απαιτούνται 67 τριμερείς διάλογοι όπως έγινε τελευταία φορά με τον κανονισμό. Επίσης, από ό,τι λένε οι προγνώμονές μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι εύχριστο ότι αποφασίσουμε, γιατί είδατε τι προβλέπει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί κανείς να προαναγγείλει ένα πολίτες. Οπότε αφού θέλετε το ένα α τότε βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια τα ανταυτά στοιχεία. Δηλαδή το Erasmus 2020 και το Connecting Europe είναι προγράμματα βέβαια τα οποία κανείς διαφωνεί την εξαίρετα θα είναι το 70% του 1α. Αλλά στην περίπτωση αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε τεράστιες περικοπές το 1α. Όπως για το πρόγραμμα Έρασμος. Άρα είναι πολύ δύσκολη η επιλογή. Ψάχνετε για αναλεκτική, αλλά όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, η δημοκρατία είναι το χειρότερο σύστημα από έχω ψάξει, αλλά τελικά εκεί καταλήγεις αφού έχεις λάβει υπόψη ό,τι άλλο υπάρχει. Οπότε, για τα κριτήρια της επιλεξιμότητας, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή ακράδαντα θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τομεακή δέσμευση χρημάτων. Γιατί το πρόγραμμα αυτό προβλέπει και αποσκοπεί στο να ελκύσουμε χρήματα ιδιωτικών επενδύσεων. Και άμα αρχίσουμε να τους περιορίζουμε, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε τον στόχο για αυτά τα 250 δις ε, επενδύσεις. Οπότε τα κριτήρια της επιλεξιμότητας θα πρέπει να είναι σχετικά απλά. Πρώτα πρώτα να υπάρχει συνέπεια με τις πολιτικές της Ένωσης, θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει δηλαδή εκείνη η λογική. Άμα δεν είναι βιώσιμο, πώς να ε, ελκύσει τους ε, ιδιώτες επενδυτές. Κατά τρίτον, να υπάρχει αυτή η προσθετικότητα. Δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει ακόμα μια φορά τα ίδια πράγματα. Ούτε θέλουμε να αποθήσουμε τους ε, ιδιώτες επενδυτές υπάρχει χρηματοδότηση όπως πρέπει. Με εγγύηση της ΕΤΕΚ. Και να μπορούμε να κινητοποιήσουμε έτσι τους επενδυτές. Τώρα το καθόδες ζήτημα των ευθυντήριων γραμμών για τις επενδύσεις εν γέννη για τις κατευθυντικές πράξεις αυτά πιστεύουμε και προκειμένου λέμε προσοχή γιατί γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη, αλλά και από το Κοινοβούλιο, όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των καθεντήριων γραμμών. Και με την της πράξη τι θα γίνει. Τα έχουμε παρατηρήσει από τα 28 κράτη-μέλη, τις 12 επιτροπές που έχετε εδώ και φαντάζεστε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θα καταλήξουμε μετά από ένα χρόνο συζήτησης να έχουμε μπροστά μας ένα χαρτοβασίλειο να διεκπαιρεώσουμε ενώ θέλουμε να υπάρχει ταχεία πρόοδος. Γιατί και με το Swiss Life πολλές φορές έχουμε πάρα πολλά μέσα τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά θεωρητικά αλλά τα αποτελέσματα είναι κάκιστα γιατί οι προϋποθέσεις της εφαρμογής ήταν πάρα πολύ περιοριστικές. Επίσης, τεχνική αρρωγή Οπότε δεν αρκεί πρικοδότηση για την τεχνική αρρωγή. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτό είναι επιπλέον του που σου Και αυτός ο κόμβος θα είναι μοναδικό σημείο πρόσβασης, αλλά επίσης θα έχουμε και όλη την άλλη ε, τεχνική βοήθεια που ήδη ε, προβλέπεται για το Horizon 2020, Connecting Europe κλπ. Μιλούμε άρα για 450 εκατομμύρια που θα πρικοδοτούν αυτή τη βοήθεια. Και μιλάμε για 20 εκατομμύρια ετησίω που είναι κάτι σαν επιπλέον. Εκεί που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τωρινά, όπω για το Είπαμε για 20 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά χρειάζονται τα ταμεία να επιστατευτούν για αυτά τα project. Υπάρχουν και project όπου δεν χρειάζεται να επιστατευτούν τα διευθυντικά ταμεία. Για τις ΜΜΕ είπατε ότι χρειάζεται και εκεί να διατεθούν κάποιοι πόροι. Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη αυτό στις προτάσεις μας. Να σας πω ότι μόνο για αυτές τις περιπτώσεις έχουμε διαθέσει ποσά στις προτάσεις μας. Πέντε δις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για μικροεπιχειρήσεις και έψιλον. Τα έξω 5 εκατομμύρια θα οδηγήσουν σε 75 δις επενδύσεων για τις ΜΜΕ που είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Επίσης είπατε ότι έχουμε το COSME, Horizon 2020, έχουν πολλά μέσα πολιτικής. Και εδώ θα έχουμε πλήρη εφαρμογή αυτών των μέσων το 2020 και για το κόσμο και για το ρίζον 2020 επομένως, οπότε θα υπάρχει και η μόγλευση η οποία αμέσως θα είναι προσβάσιμη από πλευρά των ΜΜΕ. Επίσης θα πρέπει να εμπλακούν εδώ και οι τοπικές αρχές που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για projects στη, στο Ταμείο Επενδύσεων. Όποιος θέλει. Και οι ιδιώτες μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε υπάρχει χρηματοδότηση αλλιώ και άρα είναι καλοδεχούμενοι οι τοπικές αρχές να εμπλακούν. Αλλά βέβαια να κλείσω ευχαριστώντα εισηγητής και όδης εισηγητές και την επιτροπή σας. Πιέζει πολύ ο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι με καλή διάθεση θα τα καταφέρω. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι α, θα εγώ εγώ σε αυτές τις ε, σημαντικές προτάσεις. Αλλά μα μας είπατε και ποια είναι τα όρια της δημοκρατίας. Μα εδώ όμως εμείς έχουμε εκλεγεί ε, από δημοκρατικές εκλογές, οπότε δεν θα πρέπει εδώ να τα λέμε αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι θεμητό να λέτε τις απόψεις. Η εισηγήτρια τώρα. Ευχαριστώ. και όπως είπα και στην εισαγωγή μου και σήμερα αλλά και προηγουμένως, από το 90% των ε, παρεμβάσεων πρόκειψε μία σύμπνοια. Πολύ θετικό αυτό. Και θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη για την ακαμψία που δείχνει και την αδιαλαξία της ε, σε ό,τι αφορά το χρηματοδοτικό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι εξίσου παράνομο από τη σκοπιά της Κομισιόν να πιστεύει ότι μπορεί να αφαιρέσει κονδύλια από το συνδέοντα στην Ευρώπη και το ορίζοντα 2020 χωρίς να περάσει την τακτική ετήσια ε, διαδικασία του προϋπολογισμού. Και το είπαν και οι συνάδελφοι. Είχαμε εκτενέστατες συζητήσει με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε λεπτομέρεια του συνδέοντο στην Ευρώπη και το ορίζοντα 2020. Και τώρα με μία μόνο κοντιλιά θέλετε να αλλάξετε μία τόσο εύθραυστη ε, ισορροπία και συμφωνία που είχαμε στο παρελθόν. Αμφίβολο το βλέπω. Οπότε ως προς την παρανομία ούτε και εσείς μπορείτε να ε, είστε τελείως καθαροί από αυτή την άποψη. Αντιλαμβάνομαι κάποια επιχειρήματα, τώρα δεν μπορώ να επισέλθω σε όλε τι λεπτομέρειε. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα βοηθήσει για να βρούμε σωστή λύση. Γιατί είμαστε πολύ διαλλακτικοί, ανοιχτοί να βρούμε λύσει, αλλά δεν θα είμαστε εύκολοι στι διαπραγματεύσει ε, ενδοτικοί για το συνδέοντα στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Και δεν είναι αυτή η ιδέα ή το καπρίτσιο τη ηγήτρια ή μερικών σχεδόν εισηγητών ή σε μερικών συναδέλφων σε επιτροπέ. Αυτή είναι διακομματική, ευρεία συνένεση και έχουμε πλούσια εμπειρογνωμοσία που μας στηρίζει σε αυτή τη θέση. Γιατί έχουμε εμπειρογνώμονες και ειδικού που μας βοηθούν στο έργο μας. Και ένα ακόμη θέμα που προέκυψε από πολλές παρεμβάσεις. Το θέμα της διακυβέρνησης ε, και το συναφές θέμα του earmarking, ε, των κονδυλίων ειδικού σκοπού. Γιατί θέλουμε κονδύλια ειδικού προορισμού, γιατί δεν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη τι θα συμβεί αν πρικοδοτήσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Οπότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε τις μέρες που μας έρχονται και όπως είπε ο κύριος Σέλερ να έχουμε σαφή και στεναρή γραμμή για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε καλύτερη οριοθέτηση των κριτήριων επιλεξιμότητας, όχι μόνο στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οριοθέτηση σε ό,τι έχει σχέση με τη μετάβαση της οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε διαφορετικό ενεργειακό σύστημα από αυτό που έχουμε σήμερα. Χρειαζόμαστε ψηφιακή οικονομία, τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες και θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε στα κριτήρια επιλεξιμότητας και θέλουμε ε, ε, κονδύλια ειδικού σκοπού, η αρμάκιν, γιατί στο παρελθόν δεν ήταν αρκετά αυτά που έγιναν ούτε για την ενεργειακή απόδοση, ούτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και προσβλέπουμε σε μια καλή συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά, με πλήρη στήριξη από την Επιτροπή Ήτρε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να ζητήσω αναβολή τη ψηφοφορία για να εξασφαλίσω λίγο χρόνο επιπλέον, αλλά είμαι πρόθυμη να επιταχύνω τις εργασίες και να μην αναζητήσω αναβολή. Γιατί αν ψηφίσουμε στι 14 και είναι καλό το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία και η υπερκομματική στήριξη, θα έχουμε πολύ καλό επιχείρημα για να παρεύουμε στις συμβαστικές τροπολογίες στις Επιτροπές Εκών και Προπολογισμών για τα θέματα της διακυβέρνησης, για το άρθρο 8, όχι φυσικά για τις δικές τους αποκλειστικές αρμοδιότητες. Εκεί μπορούμε, αν έχουμε ήδη εμείς ψηφίσει, να επηρεάσουμε κάπω την έκβαση ε, των συμβιβαστικών τροπολογιών στις Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμών. Στο επόμενο μισάωρο έχουμε και άλλη έκθεση. Ευχαριστώ Κάθλιν. Χειροκροτώ και εγώ. 14 του μηνός θα ψηφίσουμε, οπότε οι επόμενες εβδομάδες είναι απαραίτητες και σημαντικές και στις 20 θα ψηφίσει η Επιτροπή Έκων και Προϋπολογισμών. Καλό θα ήταν εμείς να ετοιμαστούμε πριν. Και σήμερα θα έχουμε το απόγευμα τον Επίτροπο Κανιέτε και επίσης θα έχουμε κοινή δημόσια κρόση των Επιτροπών Ήτρε, Τραν και Γιούρι για την αναθεώρηση, την ανάγκη αναθεώρησης της θερινής ώρας. Ελπίζω να δώσετε παρουσία και το απόγευμα σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση που θα έχουμε. Ευχαριστώ και ραντεβού το απόγευμα παρουσία για το Επιτρόπο Κανιέτη.